Η επόμενη σύνοδος Ολομελίας θα γίνει αύριο στις ε, Τετάρτη από τις 9 ε, μέχρι τις 1 και στη συνέχεια από το μεσημέρι τις 3 μέχρι τις 12 το βράδυ.